Οι εκθέσεις οι οποίες ε, αποτελούν και εντολή για αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της ε, συνεδρίασης. Βάσει του άρθρου 69 γ, παράγραφος 2, ένας αριθμός ευρωβουλευτών ενός ή περισσότερες πολιτικών ομάδων που ε, αντιστοιχούν στο μέσο όρο μπορεί να ζητήσουν γραπτός ε, μέχρι αύριο 3η 14 ε, Μαρτίου στις 12 το βράδυ να ξεκινήσει η ψηφοφορία για τις διαπραγματεύσεις αυτής. Εάν δεν υπάρξει έτοιμα βάση της προθεσμίας, τότε οι επιτροπές μπορούν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι την Τετάρτη μαζί με